Ladies Κυρίες ε, και κύριοι, να ξεκινήσουμε τώρα την ε, έκτακτη κοινή μας συνεδρίαση. Έχουμε ειδικού προσκεκλημένους εδώ σήμερα. Θα μιλήσω στα φιλανδικά. Οπότε, πιθανότητα, θα πρέπει να, να βάλετε τα ακουστικά σας naiset kollegat. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τιμή μου να συμπροεδρεύω μαζί με τον συνάδελφο David McAllister της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για την ετήσια συνεδρίαση που κάνουμε κάθε χρόνο με τους βραβευθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, επίσης ε, είναι εδώ ε, παρόν και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΕ του Μαρακές για την διάσκεψη του Μαρακές. Θα ήθελα να καλωσορίσω την εκπρόσωπο του κυρίου Όλεγκ Σεντσόφ, την ε, Νατάλια Κάπλαν, ε, την ξαδέρφη του, τον δικηγόρο του, τον κύριο Δημήτρη Λίντσε, ο οποίος ε, επίσης είχε προσκληθεί, όμως λόγω προβλημάτων με την πτήση του δεν μπόρεσε να παρευρεθεί απόψε. Επίσης, χαίρομαι που βλέπω στην αίθουσα δύο άλλους υποψηφίους ε, για το βραβείο Σαχάροφ. Νασέρ Ζεψάφη που εκπροσωπείται και από τους γονείς του και τους εκπροσώπους της ΜΚΟ που βοηθούν τους μετανάστες στη Μεσόγειο και σώζουν ζωές. Αυτή τη συνεδρίαση την υλοποιούμε μαζί με τις ε, αντιπροσωπείες ε, που έχουν αναμειχθεί στην απονομή του βραβείου. Καταρχήν την Κοινοφιλευτική Επιτροπή Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πρόεδρο Ντάριο Σοζάτη και τον πρόεδρο τη Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τμαρκάρα. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ε, απονείμει από το 1988 το βραβείο Ζαχάροφ σε οργανώσεις ή σε άτομα που με τις δράσεις τους ε, και τις μαρτυρίες τους και τις σκέψεις τους μας υπενθύμησαν πόσο σημαντικό είναι για τη δημοκρατική ζωή μιας χώρας ε, να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Με το πέρασμα των ετών, αυτό το βραβείο έχει γίνει μία από τι πιο συγκεκριμένε εκφράσει τη συλλογική μα δέσμευση για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη υποστήριξή μα σε όσου αγωνίζονται για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο. εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο όπου ομάδες και άτομα συνεχίζουν καθημερινά να αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη δυνατότητα να καθορίζουν τη δική τους ζωή και το μέλλον τους. Αυτός ο συνεχής αγώνας ε, μας δείχνει ε, πόσο σημαντικό είναι το όλο πλαίσιο και πόσο εύκολα μπορεί ε, να κατασταλεί σε δύσκολους καιρούς, από τη μία κρίση στην άλλη, από την υψηλή ροή των προσφύγων ε, μέχρι την τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει να μπούμε σε εμπειρασμό να θέσουμε σε κίνδυνο τα ανθρωπινά δικαιώματα που αγωνιστήκαμε τόσο να πετύχουμε απλώς στο βωμό της ασφάλειας. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι πριν δύο μήνες, ε, δύο ε, πρώην βρεβευθέντες του βραβείου Σαχάρον η Νάντια Μουράτ ε, που βρεθεί το 2016 και ο Βευρεθής ε, το 2014 τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ. Όπως είπε ο πρόεδρος Σταγιάννη, είναι τεράστια χαρά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να βλέπει να απονέμεται το βραβείο Νόμπελ ε, ειρήνη σε φέτος σε δύο βρεβεθέντες με το βραβείο Ζαχάροφ. Τώρα έχουμε πέντε βραβευθέντες με το βραβείο Σαχάροφ που στη συνέχεια έλαβαν το βραβείο Νόμπελ. Ως μέλη του Κοινοβουλίου μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό και για το έργο που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις τελευταίες δύο δεκαετίες προς ε, την υπεράσπιση των ε, υπερασπιστών των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σε αναπτυσσόμενε χώρες. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα Τιμάμε τον κύριο Όλαγκ Σέντσοφ, τον βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ και μαζί με αυτόν τιμούμε όλα τα άτομα που αγωνίζονται καθημερινά στις τοπικές τους κοινότητες ή ευρύτερα για να προσπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας τους έτσι καθολική αξία, παγκοσμία αξία. Πριν 30 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το βραβείο στον κύριο Ζαχάροφ. Τώρα, λόγω διάφορων ιστορικών συνθήκων, το βραβείο μας θα δοθεί σε έναν άλλο διαφωνούντα που είναι υποκράτηση αυτή τη στιγμή στη Ρωσία επειδή εξέφρασε δημοκρατικά τις απόψεις του με ένα εντελώς ειρηνικό μη τρόπο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο, στον κύριο Μακάλιστερ, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Thank you, Mirja, for your introductory remarks. Just a couple of words from my side as Chair of the Foreign Affairs Committee. Dear colleagues, first of all, let me underline how happy I am that the representative of our 2018 Sakharov Prize winner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 Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Όλικ, τον οποίο σήμερα εκπροσωπώ. Το βραβείο αυτό δεν θα αντικαταστήσει την ελευθερία. Η ελευθερία ξεκολουθεί να είναι πολύτιμη, πολυτιμότερη σε σχέση με οποιοδήποτε βραβείο του κόσμου. Η απεργία πείνας έχει σταματήσει problem Έχουμε ένα μικρό ζήτημα με το μικρόφωνο.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 Έχει σταματήσει την απεργία πείνας, αλλά δεν έχει αποκατασταθεί εντελώς η υγεία του ακόμη και δεν είναι και σίγουρο ότι θα επανέλθει σε μια φυσιολογική κατάσταση. Είναι στην Αρκτική, στην περιοχή Γιάμαλ, στην Τούνδρα, εκεί τάρανδη και πολικές αρκούδες ε, ε, μπορεί κανείς να συναντήσει. Εκεί τον έχουν στείλει. Έχει περάσει όλη του τη ζωή στην Κρυμαία. Και πνευμονοπάθειες και καρδιοπάθειες ε, είναι κάτι που μπορεί να το πάθουν ντόπιοι. Ο Όλεκ έχασε μαλλιά, έχασε τα δόντια του τους πρώτους μήνες της κάθριξης, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Εμένα, και όχι μόνο εμένα, με έχει εντυπωσιάσει το πόσο ενεργός είναι και πρέπει να σας πω ότι τώρα ε, βιντεοσκοπεί, ακόμα και τώρα, ε, φτιάχνει μια ταινία ε, με βάση ένα έργο ε, θεατρικό το οποίο είχε συγγράψει πριν συλληφθεί μαζί με τον κ. Νορμπάγεφ τον σκηνοθέτη ο οποίος είναι από την Κρυμαία επίσης ε, τον ε, ονομάζει αδελφό του από την Κρυμαία ε, και ουσιαστικά μεταφέρει το όραμά του, συμμετέχει στο casting και επιλέγει δηλαδή τους θοποιούς, συνεχίζει τη δουλειά του δηλαδή, συνεχίζει τον αγώνα του. Πέντε χρόνια σχεδόν έχουν περάσει, οι συνθήκες όμως επιδεινώνονται. Ο ίδιος βέβαια είναι ενθουσιώδης και ε, στηρίζει πιο πολύ αυτούς που είναι έξω από τη φυλακή, είναι ένας ήρωας πραγματικά. Και παρόλα αυτά είναι ένας απλός άνθρωπος, δεν θέλει να τον αποκαλούν ήρωα. Αυτά είχα να πω από τον Όλεγκ ένα μεγάλο ευχαριστώ για το βραβείο αυτό που του απονείματε. Ευχαριστώ. Thank you, I would like to give the to some θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιους ε, συναδέλφους ε, ε, και θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Ροζάτη, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, με την Ουκρανία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καπλάν, σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, φέτος ε, το βραβείο Ζαχάροφ απονεμήθηκε στον Όλεκ Σέντσοφ σε έναν άνθρωπο ο οποίος με την αποφασιστικότητά του να παραμείνει ελεύθερος άνθρωπος παρά μία παράνομη δίκη και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, ο άνθρωπος αυτός ενσαρκώνει την ελευθερία των αγώνα κατά της ρωσικής καταπίεσης. Είναι ήρωας, όπως πολύ σωστά είπατε, ήρωας για όλους μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έχουν στηρίξει την υποψηφιότητά του. Όπως ε, κύριε Πρόεδρε θα έχετε διαπιστώσει, ο αγώνας για την απελευθέρωση του Όλεξ και όλων των άλλων κρατουμένων που παράνομα κρατούνται από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αυτός ε, δεν είναι ο μόνος ε, λόγος γιατί αγωνιζόμαστε σήμερα. Αγωνιζόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια από τότε που υπήρξε το Φεβρουάριο του 2014 η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια σειρά από ψηφίσματα που που καταδικάζουν ε, αυτές τις επιθετικές πράξεις ε, και το Κοινοβούλιο απαιτεί την απελευθέρωση κρατουμένων από τις ε, ρωσικές φυλακές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει στο να επισημαίνει σε όλο τον κόσμο τις περιπτώσεις όλων αυτών που τολμούν να διαφωνούν με την προσάρτηση της Κρυμαίας και γι' αυτό τον λόγο κρατούνται παρότι είναι όλοι Ουκρανοί πολίτες. Έχουμε λοιπόν εκφράσει τη θέση μας σε πάρα πολλά ψηφίσματα ε, τα οποία έχουν στηριχθεί από μια συντριπτική ε, διακομματική ε, πλειοψηφία και αυτό το υπογραμμίζω. Υπάρχει μια ευρύτατη πλειοψηφία η οποία στηρίζει επίμονα την προσπάθειά μας να απελευθερωθεί ο Λεξέντσοφ από τις ρωσικές αρχές. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα το κάνουμε αυτό με κάθε ευκαιρία και θα συνεχίσουμε να το απαιτούμε και με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ουκρανία. Είμαστε πολύ δραστήριοι, προσπαθούμε να συζητάμε με τους Ουκρανούς φίλους και συνομιλητές διάφορους τρόπους για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε το στόχο μας έτσι ώστε ο Όλεξ Σένσοφ και όλοι οι συγκρατούμενοι του να αφαιθούν ελεύθεροι. Τις προηγούμενες εβδομάδες είδαμε άλλη μία απόδειξη της κοινικής συμπεριφοράς του Κρεμλίνου. Συνέλαβαν 24 Ουκρανούς διασώστες και όλοι αυτοί τώρα κρατούνται ε, σε, είναι προφυλακισμένοι σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα κοντά στη Ρωσία. Αυτό είναι άλλο είναι ένα παράδειγμα επιθετικής πολιτικής της Ρωσίας η οποία δεν διστάζει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο για να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους. Αυτήν λοιπόν την ε, εβδομάδα πρόκειται να απονείμουμε ε, το βραβείο στον Όλεξέντσοφ κατά κύριο λόγο για να αποδείξουμε ότι υποκλεινόμεθα στο θάρρος του είναι έμπνευση για όλους όσοι καταπιέζονται σε, όλα τα, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Πέρα όμως από αυτό επιθυμούμε να δράξουμε την ευκαιρία για να εντείνουμε την πίεσή μας έναντι του Κρεμλίνου, να πούμε με στεντόρια φωνή ότι εμείς ε, δεν καμπτώμεθα από την προπαγάνδα του Κρεμλίνου και γνωρίζουμε πολύ καλά το τι διαδραματίζεται και στη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι επίσης ε, η δική μας ε, φωνή να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους Ουκρανούς κρατούμενους, σε ρωσικές φυλακές, ε, οι οποίοι κρατούνται γιατί απλά αρνούνται να παραδεχθούν την ρωσική κατοχή. Εμείς στο Κοινοβούλιο δεν το ξεχνάμε αυτό, με κάθε ευκαιρία ζητάμε την απελευθέρωσή τους. Κυρία Κάπλαν, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβιβάσετε τις ευχές μας, τις θερμότατες ευχές μας στον Όλεξ Έντσοφ και να του εκφράσετε και το σεβασμό που νιώθουμε για το πρόσωπό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ροζάτη και τώρα ο Κάρας ε, για την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Herr Vorsitzender, liebe Frau Kaplan, Sie Πρόεδρε, αξιότιμε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά που ακούσαμε ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Είναι ένα πρόβλημα που περιγράψατε, ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας. Αφορά τον Όλεκ και όλους τους ανθρώπους. Ο Όλεκ ε, αποδεικνύει ότι υπάρχουν ε, αρνητικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα είναι και ένα σύμβολο για όλους τους ανθρώπους και αγωνίζεται για αυτούς. Ε, σήμερα είναι μια ειδική ε, ευκαιρία, γιατί σήμερα στις 10 ε, Δεκεμβρίου έχουμε την 70η επέτειο από την πρώτη διακήρυξη των Οικουμενικών Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σας χαιρετίζουμε ω εκπρόσωπο του Όλεξ Σας χαιρετίζουμε θερμά και χαιρετίζουμε την παρουσία σας, ειδικά αυτή την ημέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Αντιπροσωπεία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ρωσία. Η αντιπροσωπεία χαίρεται και είναι και υπερήφανη για το ότι έχουμε επιτύχει αυτή την ε, συνάντηση ε, μαζί σας ε, εσείς ε, βλέπουμε το πρόσωπό σας, σας βλέπουμε, ήρθατε εδώ, ήρθατε σε μας και με αυτή την συνάντησή μας ε, θέλουμε να τιμήσουμε το θάρρος ε, και την τόλμη του Όλεκ Σένσοφ. Δεν μπόρεσε να έρθει, δεν τον άφησαν και αυτό αφορά και τόσους άλλους Ουκρανούς πολίτες οι οποίοι μετά από άδικες δίκες βρίσκονται εγκλίστηκαν στις ρωσικές φυλακές. Αυτό είναι ιδιαίτερα επώδυνο και είναι κάτι απόλυτα κατακριτέο. Ως πρόεδρος λοιπόν αυτής της αντιπροσωπείας, εγώ με τους συναδέλφους μου προσπαθώ ε, στο πλαίσιο που μας επιτρέπεται να γύρουμε γέφυρες. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν κόκκινες γραμμές, υπάρχουν κόκκινες γραμμές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίως γι' αυτό. Και ξέρετε, οι κόκκινες γραμμές είναι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός ε, του διεθνούς δικαίου. Αυτές είναι για μας οι κόκκινες γραμμές. Αυτές ε, έχουν θεμελιώδη σημασία για το Κοινοβούλιο. Εμείς ε, έχοντας μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλλον η Ρωσία ως μόνιμο μέλος ε, του Συμβούλιο Ασφαλείας και ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών, οφείλει να νιώθει ιδιαίτερη ευθύνη έναν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς δεν θα δεχτούμε καμία παραβίαση και καμία απόκληση από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας, εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμά, ε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Στο Ντομπάς ε, συνεχίζεται η βία αντίδραση, η τήρηση των συμφωνιών του Μίνσκ ε, είναι όλο και πιο μακριά. Υπάρχει επιπρόσθετα και η επιθετική και ανεύθυνη συμπεριφορά του ρωσικού στρατού. Και αυτό έχει προκαλέσει νέες εντάσεις στη θάλασσα του Αζόφ για την σταθερότητα και την ειρήνη της Υπήρου μας η επαναφορά της εδαφικής ακαιρεότητας της Ουκρανίας είναι εκ των καθοριστική σημασίας. Μπορούμε λοιπόν να σας υποσχεθούμε σήμερα ότι θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε απερίφραστα την επιδείνωση των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Η καταπίεση των ακτιβιστών ή των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, ε, του πολιτισμού, ε, νόμιο όλο και περισσότερο ε, κομμένοι και ραμμένοι σε κάποιες ανάγκες, αυτό οδηγεί σε μία περιδίνηση, μία κοινωνική επιδίνωση της κατάστασης. Έχουμε λοιπόν ε, αυτή την ρωσική προπαγάνδα που ε, ρίχνει λάδι σε αρνητικά συναισθήματα, υποδαβλίζει αρνητικά συναισθήματα. Ο Λεξένσοφ είναι σύμβολο, σύμβολο για πολλούς που έχουν καταδικαστεί άδικα. Εμείς λοιπόν ελπίζουμε ότι ε, θα μπορούν όλοι αυτοί σύντομα να φεθούν ελεύθεροι να βγουν από τις φυλακές, ε, να μπορούν ως Ουκρανοί να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, ε, να μπορούν να εργαστούν, να ζήσουν ε, χωρίς φόβο, χωρίς να αισθάνονται την ποινική δίωξη. Οι απόψεις, οι ιδέες είναι ελεύθερες, οι ιδέες δεν μπορούν να εγκλειστούν σε φυλακές. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον Όλεκ Σέντσοφ και για όλους τους συμπολίτες του. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρεμπεκά Χάρμς, η οποία είναι πρόεδρος ε, της ε, Euronest Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Η Euronest ε, αποτελεί ένα θεσμό όπου συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με χώρες της Ανατολικής Γειτονικής Σχέσης και την Ουκρανία. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Θα μιλήσω γερμανικά, όπως και προλαλή σας. Χαίρομαι πολύ που υπάρχει τόσο μεγάλη συνένεση μεταξύ των συναντέλφων για την απονομή του φετινού βραβείου Ζαχάροφ στον Όλεξ Σεντσόφ. και νομίζω ότι αυτή η ευρεία συνένεση δείχνει επίσης ότι και τα αιτήματα τα οποία ε, υπεράσπισε με την απεργία πείνας του Όλεγ Σεντσόφ έχουν γίνει αντιληπτά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ξαδέρφη του, η Νατάλια, καλώς ήλθατε Νατάλια, είναι πολύ καλό πιστεύω εδώ και που υπογραμμίσατε ότι ο Όλεκ ήθελε να κάνει ταινίε, αλλά ήθελε να τις γυρίσει ελεύθερος και αγωνίζεται για την ελευθερία της Ουκρανικής του πατρίδας, της Κρυμαίας ε, και είναι ένας ε, φιλιρινικός ακτιβιστής. Ε, το 2014 αγωνίστηκε ειρηνικά και καταδίκασε την συμπεριφορά της Ρωσίας και την προστάτηση της Κρυμαίας και γι' αυτό φυλακίστηκε και σίγουρα έχετε και εσείς Νατάλια και άλλοι αγωνιστεί για την απελευθέρωση του Όλεγκ και ε, θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω αυτή την ε, επιθυμία και να πω ότι δεν θα παρετηθούμε ε, της ιδέας αυτής. Θέλουμε να απελευθερωθεί ο Όλεγκ και ελπίζουμε πραγματικά υπονομή του βραβείου. Αυτή η απόφαση να απονείμουμε αυτό το βραβείο στον Όλεγκ ελπίζουμε να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα τη συντομότερη δυνατότητα τη απελευθέρωσή του, την οποία θα χαιρετήσουμε εδώ. Πρέπει όμως να τονίσω ότι ο Όλεξεν Τσόφ σε καμία περίπτωση ε, δεν κινήθηκε μόνο για ε, προσωπικούς λόγους. Φυσικά θέλει να γυρίσει ταινίε, ε, αλλά ξέρουμε και άλλους δημοσιογράφους από τον Ντομπάς, από την Ουκρανία, που θέλουν να εργαστούν. Ξέρουμε αγρότες από την Κρυμαία που θέλουν και αυτοί να συνεχίσουν να εργάζονται, να ασκούν το επάγγελμά του. Είναι πάρα πολλοί οι Ουκρανοί αυτοί οι πολίτες που κρατούνται στη Ρωσία, κρατούνται στις φυλακές και πληρώνουν το ίδιο τίμημα. Με αυτό πληρώνει όλη Σεντσόφ. Ε, το είπε και το είχε επαναλάβει πολλές φορές ε, ότι και την απεργία πείνας την ε, ε, κάνει για την ελευθερία και αυτό το έκανε όχι μόνο για τον εαυτό του και για όλους όσοι έχουν χάσει την ελευθερία τους στην Κρυμαία. Σας ευχαριστούμε Νατάλια που είστε εδώ. Πρώτα, ευχαριστώ πολύ και τη Ρεμπέκα Χάρμς για τα πολύ ξεκάθαρα φιλικά λόγια και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους μου να είναι στον πιο σύντομοι για να ακούσουμε και την ευθρολή της κυρίας Καπλάν, εκ μέρους του ΕΛΚΟ Έντουαρτ Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να κρουσίσω ενθερμά την κυρία Καπλάν αλλά και τους ε, υπόλοιπους ε, φινελείς του βραβείου Σαχάροφ ε, φέτος. Χαίρομαι που συναντιόμαστε φέτος με αφορμή το βράβευση του Ολεξένσοφ, εγώ μαζί με τον Μιχαλ Γκάλερ πρότεινα τον Ολεξένσοφ ε, για την πολιτική μας ομάδα. Σήμερα είμαι περήφανος που πετύχαμε ε, με την βράβευση του και την υποψηφιότητά του και ευχαριστώ πολλούς συναδέλφους ε, για την υποστήριξη. Η υποψηφιότητα του Ολεξένσοφ βασίστηκε στην αντίστασή του στη ρωσική κατοχή στην Κρυμαία και στον αγώνα του για τους πολιτικούς κρατουμένους ε, στη Ρωσία. Ο Όλεγ Σέντσοφ στις πεπιθήσεις του ήταν κάθετος, μόνος του στάθηκε κατά της αδικίας και του συστήματος που ήθελε να τον ποινικοποιήσει. Μας έδειξε πόσο έτοιμος είναι να θυσιάσει, πόσο είναι να πώ έτοιμο ε, να ε, αυτό όταν έκανε 145 μέρε απεργία πείνα. Ο Όλεκ αποφάσισε να κάνει αυτή την ε, ριζοσπαστική έκκληση, ελπίζοντας να ακουστεί η φωνή του και ότι έτσι θα διαδώσει οι αξίες που αφορούν την ελευθερία, την αλήθεια και τη δημοκρατία. Ακούσαμε την έκκλησή του και είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τη φωνή του. Η έκκλησή του τον καθιστά ε, κρατούμενο συνείδησης ε, που αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης και καθώς ε, πιστεύουμε στην υπεροχή αυτών των αξιών ε, κατά ε, της σκληρής βίας, πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή με την υποψηφιότητά του για το βραβείο Ζαχάρου Φόλεξ Σέντσοφ. είναι ένας αθώος άνθρωπος που είναι ακόμη στη φυλακή. Δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σιωπηλοί. θα πρέπει να σεβόμαστε το κράτος δικαίου, την ελευθερία της σκέψης, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να συμπενθυμίσω ότι η ελευθερία της σκέψης είναι ο χειρότερος εφιάλτης για όλα τα ε, δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα, ε, καθώς δεν τους επιτρέπει να ελέγχουν ε, τους ανθρώπους. Ε, πρόκειται για ένα ισχυρό όπλο εναντίον τους. Δεν θα πρέπει να πεθάνουν στη σιωπή η ελευθερία και η ελπίδα. Ως κάποιος που προέρχεται από την πρώην Τσεχοσλοβακία, για πάνω από 20 χρόνια είχαμε σοβιετικά στρατεύματα στην επικρατεία μας και θεωρώ την ε, βράβευση του Όλεκ Σένσοβ μια αναγνώριση όλων ε, των φωνών που δεν δίστασαν ε, να εξεγερθούν κατά της ειδικίας. Όλες αυτές οι φωνές πρέπει να ακουστούν. Παρ' όλα αυτά, έχω μεικτά συναισθήματα σήμερα, καθώ το όνομα του Αλεξέντσοφ ε, θα εμφανιστεί στο κατάλογο των βραβευθέντων μα με το βραβείο Σαχάροφ για την ελευθερία τη σκέψη. Και αυτό ο ίδιο εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή ε, στη Ρωσία και η υγεία του είναι σε εύθραστη κατάσταση. Όταν υποβάλαμε την υποψηφιότητά του, είχα μια μικρή ελπίδα ότι θα είχα την ευκαιρία να το συναντήσω προσωπικά κατά τη διάρκεια τη τελετή ε, απονομή. Δυστυχώ δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα ε, να του πω να παραμείνει ισχυρός ε, στις πεπιθήσεις του γιατί δεν είναι μόνος του στον αγώνα του κατά της αδικίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. <clears throat> Κύριε Κούκαν, και θα ήθελα να πω σε εσά κύριε Καπλάνο ότι ο κύριος Κούκαν την προηγούμενη εβδομάδα ε, έκανε ένα ντοκιμαντέρ για την δίκη, ε, για την ταινία «Δίκη», ε, παραβρέθηκα κι εγώ και αυτό ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είμαστε ένα πολυσχηδέ κοινοβούλιο. Έχουμε οκτώ πολιτικέ ομάδες. Θα δώσω λοιπόν το λόγο σε κάθε ένα εκπρόσωπο από αυτές τι πολιτικέ ομάδε. Επόμενη είναι οι σοσιαλδημοκράτε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσά, κυρία Νατάλια Καπλάν. Ε, που είστε οι εξαδέλφοι του κυρίου Όλεξ Σέντσοφ. Ε, θέλω να σας πω ότι είναι τιμή για μας το να σας βλέπουμε σήμερα εδώ. Ε, εγώ, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, θα ήθελα να καλωσορίσω και τους ε, δύο άλλους υποψήφιους, τους εκπροσώπους των Saving Lives που έσωσαν πολλές ζωές στη Μεσόγειο και τους εκπροσώπους ε, τους άλλη ομάδα, ε, οι οποίοι και αυτοί επέδειξαν θάρρος και ειλικρινή ε, στράτευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επέδειξαν και πνεύμα αλληλεγγύης. Ο Όλεκ Σέντσοφ, συγγραφέας κινηματογραφιστής, ε, πολιτικός ακτιβιστής, ε, ο οποίος ε, χρησιμοποίησε ειρηνικά την τέχνη του για να εκφράσει την αντίθεσή του, να ασκήσει κριτική στην Ρωσία και στην παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. Στυλίτεψε τις παράνομες ε, πράξεις κατά των Τατάρων της Κρυμαίας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλο και εμάς εκπροσωπεί το θάρρος, την αποφασιστικότητα και βέβαια και τον αγώνα κατά της ε, καταποίησης, τον αγώνα υπέρ της ελευθερίας έκφρασης. Με βάση την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ελευθερία της έκφρασης είναι αναφέρετο δικαίωμα για κάθε άνθρωπο. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία παρέμβαση να μην υπάρχουν παρεμβάσεις από μέσα ενημέρωση και αυτό ανεξάρτητα από σύνορα. Ε, ο μη σεβασμό όμως αυτής της ελεύθερης έκφρασης είναι εκείνος που οδήγησε τον όλευ στις φυλακές. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλους αυτούς τους ταραλέους ανθρώπους, τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες, τους κινηματογραφιστέ τους φωτογράφους, τους αμύντορες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους απλούς ανθρώπους για να καταθέτουν για ε, καταχρήσεις εις βάρος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προστατεύουν την δημοκρατία, γιατί όλο και περισσότερα διακυβεύονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι το βραβείο ε, Ζαχάροφ θα είναι κάτι που θα ξυπνήσει την ρωσική κυβέρνηση και θα την οδηγήσει στο να αφήσει ελεύθερο τον Όλεγκ και τους άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους ε, που κρατούνται σε φυλακές ε, της Ρωσίας. Θα ήθελα να παραθέσω από τον Όργουελ που είπε ότι αν η ελευθερία σημαίνει κάτι, τότε αυτό το κάτι είναι το δικαίωμα να λέει κανείς ανθρώπους αυτό που δεν τους αρέσει να ακούν. Εκ μέρους λοιπόν της δικής μου της πολιτικής ομάδας, κυρία Κάπλαν, θα θέλαμε να διαβιβάσετε την αμέριστη υποστήριξή μας τις καλύτερες ευχές μας ε, στον εξάδελφό σας ε, να συνεχίσει τον αγώνα του για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές της Ρωσίας. Ευχαριστώ, Πόστ, Κυρία Πόστ, δεν υπάρχει κουράσπος εδώ από το ECR. Α, εκεί. Συγγνώμη, τόσο μακριά προς τα δεξιά δεν κοιτάζω ποτέ. Συγγνώμη, καθυστέρησα κι εγώ. Κάθισε εδώ στη γωνία. Θα ήθελα να μιλήσω Ολλανδικά. Εγώ μπορώ να πω ότι και το ECR υποστήριξε ξεκάθαρα την υποψηφιότητα του Όλεγκ Σέντσοφ, καθώς πάντοτε υποστηρίζαμε την Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στον αγώνα για την αναξαρτησία της και την ε, εδαφική ακαιρεότητά της. Κανένα ε, λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων, επειδή εκφράζει απλώ κάποιε σκέψει, δεν μπορεί να καταλήξει στην φυλακή. Σίγουρα αυτό γίνεται βάσει ενός αθρού κατηγορητηρίου. Εμείς ανησυχούμε για την υγεία του Όλεγκ Σέντσοφ Ξέρουμε ότι δεν συμμετείχε σε αυτές τις ε, ενέργειες ε, που το καταλογίζουν Είναι σημαντική η απονομή του βραβείου αυτού και για όλους τους άλλους πολιτικούς κρατουμένους στη Ρωσία. Σημαίνει ότι εμείς συνεχίζουμε με δυνατή φωνή να λέμε ότι δεν ξεχνάμε το Σέντσοφ ούτε τους υπόλοιπους πολιτικούς κρατουμένους της, ε, τους Ουκρανούς. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που δίνεται από αυτό το κοινοβούλιο μια στιγμή χρονική, οπότε βλέπουμε παντού αυταρχικές τάσεις παγκοσμίω σε ό,τι μας αφορά να διαβιβάσετε τα χαιρετίσματά μας ε, στον Όλεγκ Σέντσοφ καθώς ε, και τις καλύτερες ευχές μας. Ευχόμαστε να απελευθερωθεί σύντομα από αυτή την άδικη φυλάκιση. Σας ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε... στους ε, φιλελεύθερους στο Κοινοβούλιο. κ. Σιλαβίτσιος. Πρόεδρη αγαπητή Νατάλια, ε, αγαπητοί υποψήφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, το φετινό βραβείο Ζαχάροφ ε, είναι σοκαριστικά συμβολικό. Αυτά τα σύμβολα λένε πολλά για το πόσο σοβαρός και δυνηρός είναι ο αγώνας ε, για την ελευθερία και τα δικαιώματα αλλά και σήμερα όπως και στη Σοβιετική εποχή. Ε, ακριβώς πριν 30 χρόνια, το 1988, το πρώτο βραβείο Ζαχάροφ απονεμήθηκε στον Έλσον Μαντέλο και στον Ανατόλη Μαρτσένκο. Μετά το θάνατό του ε, και συνάδελφος ε, συμμετείχε σε αυτή την ε, ε, απονομή. Πριν 30 χρόνια ο Ανατόλη Μάντσοκ είχε ιδρύσει το, την ομάδα Ελσίνκη είχε αναγνωριστεί ως υπερθυμόν ένα πολιτικός κρατούμενος ε, στην Σοβιετική Ένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αντρόη Σαχαρόφ, ο Μάντσερκο ήταν ο πρώτος που μίλησε και έγραψε για ε, φυλακές ε, και γκούλακ μετά τη στελινική εποχή. Γι' αυτό πέρασε 20 χρόνια σε σοβιετικές ε, φυλακές και απελάθηκε στη Σιβηρία. 20 χρόνια. σε δύο μέρες θα ε, ε, απονέμουμε το βραβείο στον Αλεξένσοφ ε, που κρατείται στη Ρωσία του Πούτιν. Δεν θα είναι ο πρώτος, αλλά ευτυχώς είναι ζωντανό σε αντίθεση με το Μάρτσενκο. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό σε αυτός ο συσχετισμός ε, μεταξύ της ε, μετασταλινικής Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας του Πούτιν είναι κάτι σοκαριστικό. Ο Όλεγκ έχει δείξει μεγάλο θάρρος, ε, είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος και ένας ελεύθερος πολίτης, ο οποίος υπερασπίζεται δημοκρατικά ιδεώδη και τη δημοκρατία και την ελευθερία, καταρχήν στο Μαϊντάν και κατόπιν στην Κρυμαία, στην πατρίδα του και ο οποίος συνεχίζει τον αγώνα του ακόμη και μέσα από τη φυλακή, όπως μας είπε η Νατάλια και αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αγωνίζεται εκ μέρους όλων των Ουκρανών πολιτικών κρατομένων ε, που έχουν ε, φυλακιστεί από το καθεστώς του Πούτιν σε πολύ εχθρικό περιβάλλον. Όπως και στη μετασταλινική εποχή, φαίνεται ότι το τίμημα για την αμπρομή του βραβείου Ζαχάροφ να είναι 20 χρόνια στην Βόρεια Σιβηρία. Είμαι βέβαιος ότι αυτός ο συμβολισμός προσθέθηκε στην ε, υπόθεση ε, του Αλεξάντσοφ στο Κρεμλίνο με ένα πολύ κοινικό μήνυμα ε, να κρύβεται από πίσω. Κυρίες και κύριοι, ο Όλεξέντσοφ αποτελεί ένα σύμβολο ενός αγώνα αυτοθυσίας κατά του σοβινισμού και της επίθεσης στον 21ο αιώνα, κατά της προσάρτησης και της κατοχής. Και αγωνίζεται για δικαιώματα και ελευθερίες που περιλαμβάνονται στην ε, Οικουμενική Διακήρυξη των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ελπίζω ότι το παράδειγμά του θα δώσει μία ενθάρρυνση που χρειάζεται για τους ε, ανθρώπους που αγαπούν την ελευθερία στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κρυμαία. Επίσης, ελπίζω ότι θα μας ενθαρρύνει Εμά, του πολιτικού που εκπροσωπούμε τον ελεύθερο κόσμο να μην κάνουμε συμβασμού στην υπεράσπιση τη ελευθερία και τη δικαιοσύνη και να σταματούμε καθεστώτα όπω αυτό στο Κρεμπλίνο. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τη μοίρα του Όλεκ στη φυλακή, να ζητήσουμε άμεση απελευθέρωση 70 πολιτικών κρατουμένων και 24 ε, ναυτικών ε, Ουκρανών ε, που πρόσφατα εγμαλωτίστηκαν στην ε, ε, περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Ελπίζω ότι θα έρθει ο καιρός που θα απελευθερωθεί όλο και θα μπορέσουμε να τον χαιρετήσουμε εδώ, σε αυτόν τον οίκο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Petras. Σε ευχαριστώ, Πέτρας. Εκπρόσωπος ε, των Πρασίνων, θα ήθελατε το λόγο, παρακαλώ. Σας ε, καλωσορίζουμε κυρία Καπλάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν τον γνωρίζω τον Όλεξ Έντσοφ. Ε, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να πάω στην Ουκρανία. Όμως πρέπει να σας πω ότι με εντυπωσιάζει πάρα πολύ το ότι όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έγκριση φυλακές και νιώθουν όλη αυτή την πίεση, παρόλα αυτά συνεχίζουν τον αγώνα τους για αυτούς που είναι έξω από τις φυλακές. Βλέπουν τα, το άδικο ε, που συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους και δεν έχουν κατά νου μόνο το δικό τους τον πόνο. Έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή ε, που χαρακτηρίζεται από όλο και μεγαλύτερη αστάθεια. Έχουμε δικτατορικά καθεστώτα, τα οποία ε, μάλιστα κατά περίπου τρόπο αναλαμβάνουν την κυβέρνηση και με δημοκρατικές ε, διαδικασίες και πολλές φορές πάλι όχι. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που ακολουθούν τον δικό τους δρόμο. Το δρόμο της ελευθερίας, της δημοκρατίας και δεν δέχονται να τους αφαιρέσει κανείς το δικαίωμα να λένε αυτό που κατά τη γνώμη τους είναι είναι το σωστό και αγωνίζονται ειρηνικά για τις πεπιθήσεις τους. Εγώ λοιπόν εδώ και 4,5 χρόνια βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και κάθε φορά ήταν πολύ δύσκολο να επιλέξει κανείς ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους για βραβείο Ζαχάροφ. Εγώ νομίζω όλοι το αξίζουν, πάντα όλοι όσοι προτάθηκαν και μένα με ενθαρρύνει το γεγονός ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, δεν ε, τοούνται ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από το στρατό, συνεχίζουν τον δρόμο τους. Αυτό λοιπόν είναι πολύ θαραλέο. Μας δίνει θάρρος και ελπίδες για τη δημοκρατία μας και για το μέλλον. Εύχομαι ο Όλεκ να μπορεί να υπολογίσει κάπως πότε θα βγει από τη φυλακή. Εύχομαι ολόψυχα να ε, αναρωσεί να νιώθει καλύτερα και σε όλους τους άλλους που βρίσκονται στον κατάλογο των υποψηφίων, σε όλους αυτούς εύχομαι να έχουν το θάρρος και την αισιοδοξία να συνεχίσουν απαρασάλευτα το δρόμο τους. Γιατί ε, είναι δύσκολο, αλλά υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για το ίδιο όφελος, αλλά προσπαθούν να επιτύχουν κάτι το καλό γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Χαιρετίσματα, πολλά χαιρετίσματα στον όλο και ελπίζω να τα ξεπεράσει όλα χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητή συνάδελφο. Η Γκουε δεν είναι παρούσα, ούτε η ομάδα η FDT. Δεν ξέρω αν, ούτε και το εθνικό μέτωπο, ε, δεν ξέρω αν κάποιος ε, θέλει το λόγο. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλα και μετά η κυρία Καπλάν μπορεί να ολοκληρώσει. Ο κύριος Γκάλα, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Σας καλωσορίζω θερμά και σας και τους ε, εκπροσώπους ε, των δεύτερων και τρίτων υποψηφίων. Ε, συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, δεν θέλουν να τα επαναλάβω. Μόνο δύο-τρεις ερωτήσεις έχω να κάνω. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λιγάκι πώς ακριβώς το έμαθε ο Λεξένσοφ ότι κέρδισε το βραβείο. Αυτό είναι το ένα που με ενδιαφέρει. Και το δεύτερο, ε, στον, ε, ε, στη φυλακή που βρίσκεται από τότε που το απονεμήθηκε το βραβείο, τι έγινε, του φέρονται καλύτερα, χειρότερα, οι άλλοι συγκρατούμενοι ξέρουν, έμαθαν ότι κέρδισε το βραβείο. Έχει δημιουργηθεί αλληλεγγύη ανάμεσά τους. Και μία τρίτη ερώτηση η ρωσική κοινή γνώμη, οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι ακριβώς κάνουν με την περίπτωση του Σένσοφ. Συζητιέται το θέμα αυτό ανάμεσα στους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν ε, κάποιες ε, πρωτοβουλίες ε, για να απαιτηθεί από την κυβέρνηση η απελευθέρωσή τους. Είσαστε μόνοι σας. Ξέρω ότι η Ουκρανία είναι ένα θέμα, αλλά το θέμα που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι πώς ακριβώς ασκείται πίεση στη Ρωσία και επίση να μας πείτε τι ακριβώς ε, περιμένετε εσείς από τις δικές μας κυβερνήσεις σε σχέση με τον Ένσοφα. Αυτές οι ερωτήσεις είχα να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκάλα για τις ακριβείς ερωτήσεις. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Κυρία Καπλάν, ακούσατε τι ρώτησαν οι συνάδελφοι. Οι ερωτήσεις ήταν και πολύ συγκεκριμένε. Ε, Χαίρομαστε που θα σας ακούσουμε. Μπορείτε να μιλήσετε όσο θέλετε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά την υγεία του όλοι ναι, αναρώνει. Ε, τον τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί η υγεία του, όπως είπατε και εσείς, αλλά όταν σταμάτησε την απεργία πίνας άρχισε κάπως να βελτιώνεται. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν τον επισκέπτονται ανεξάρτητοι ιατροί τον Όλεγκ. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με τα βεβαιότητα πώς έχει κατάσταση της υγείας του, διότι δεν, λάβουμε, δεν λαμβάνουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι. Ότι μας λένε οι γιατροί της φυλακής ε, ακούμε και από τον ίδιο τον Όλεγκ. Και όλα αυτά είναι ανησυχητικά σε ό,τι τώρα αφορά την ε, ε, θεραπεία του. υπάρχει ένας νόμος στη Ρωσία μπορούσες να στέλνεις δέμα 20 ε, ε, κιλά. Εμείς στείλαμε ένα τέτοιο δέμα, ε, επειδή όμως αυτοί μας είπαν ότι ήταν πιο βαρύ, δεν του το έδωσαν. Εκεί όμως υπήρχαν όλα τα απαραίτητα για να επιβιώσει ζεστές κάλτσες, αποξηραμένα φρούτα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Άρα δεν μπορούσαμε να του παραδώσουμε αυτό το δέμα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Αλλά αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Ο ίδιος βέβαια ίσως έχει συνηθίσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην καθημερινότητά του. Σε ό,τι αφορά όμω ε, του Ρώσου υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ναι, υπάρχουν ε, στην ε, Ρωσία. Δεν ξέρω πώ έχουν καταφέρει να επιβιώσουν στην Ρωσία, γιατί και εγώ Ρωσίδα επίκοση. Μα απλά εγκατέλειψα τη Ρωσία πριν από δύο χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο για αυτού να συνεχίσουν το έργο του στη Ρωσία. Και αυτό όχι απλά και μόνο γιατί υποστηρίζουν την Ουκρανία. Δεν υποστηρίζουν τα δικαιώματα μόνο των κρατών, αλλά όλων των πολιτικών κρατουμένων. Γιατί στη Ρωσία κρατούνται και Ρώσοι και άλλοι αντιφρονούνται εθνικότητες, άλλων ε, εθνικότητων και άνθρωποι που ζητούν ε, παραδείγματος ανταλλαγή των κρατουμένων ε, από την κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η τάση, αλλά σε ό,τι αφορά μαζικές διαδηλώσεις αυτό είναι αδύνατον να γίνει, διότι αν κάποιο κατεβεί στον δρόμο να διαδηλώσει, θα μπει φυλακή. Δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όμω ε, συνεχίζουν να αγωνίζονται. Για παράδειγμα, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρει αυτό το δέμα ο Όλεγκ. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν, αν φανταστεί κανεί και πώ ζει, σε τι συνθήκε ζει στη φυλακή. Οι ελπίδες μου δεν έχουν ε, πεθάνει, γιατί ε, ε, αυτό δεν θα είχε κανένα νόημα. Ελπίζω να βρεθεί και να μπορέσει να ασκηθεί πίεση στο Τσάρο να πιστεί ότι δεν είναι η καλή επιλογή ε, να ε, παραμένει στη φυλακή στα σίδερα ο πραγματικά καταπονήθηκε με την ε, απεργία πείνας, αλλά ε, ουσιαστικά ε, είχε ένα πάρα πολύ ισχυρό στόχο, την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Ο αγώνας του, η απεργία πείνας του ήταν για όλους, όχι για τον εαυτό του μόνο αλλά για όλους τους κράτους πολιτικούς κρατουμένους. Αυτό ήθελε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ερωτήσεις, σχόλια έχετε κάποιος, ίσως. Όχι από ό,τι βλέπω. Τότε να δώσω το λόγο στον Κρίστιαν Πρέντα, από την ιδιότητά του ως αντιπροέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντικαστά τον κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να κάνω το κλείσιμο αυτή τη συνεδρίαση που διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ανάπτυξη και την Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Μαζί με την υποστήριξη της ε, αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Ουκρανία και την αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτική Συνεργασία. Δουλεύει το σύστημα. Ε, ε, και την Επιτροπή λοιπόν Κοινοβουλευτική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία. Δύο λόγια από πλευρά μου να πω ότι γιορτάζουμε και τα 70 χρόνια ε, της ε, Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα σήμερα είναι η επέτειος 10 ε, Δεκεμβρίου. Εδώ στο Κοινοβουλίο οργανώσαμε μια εβδομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να προετοιμάσουμε την ημέρα αυτή. Και επειδή βρισκόμαστε 70 χρόνια μετά, θα πρέπει να υπενθυμίσω τον ε, την παγκόσμια εμβέλεια αυτής της ε, διακήρυξης. Ε, συχνά λέγεται ότι η διακήρυξη αυτή αφορά μόνο την Ευρώπη και μάλιστα ένα μέρος της Ευρώπης. Και λένε ότι δεν μας αφορά η διακήρυξη αυτή. Γι' αυτό ε, θέλουμε σε άλλες γεωγραφικές περιοχές να υιοθετήσουμε άλλες πιο περιορισμένες διακήρυξεις. Όμως πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η διακήρυξη αυτή είναι παγκόσμια, είναι οικουμενική, γιατί τα δικαιώματα είναι ε, ουσιαστικά οικουμενικά. Δεν αφορούν μόνο ένα λαό και μια κοινωνία. Επίσης, να σας υπενθυμίσω ένα πολύ λυπηρό γεγονός που έλαβε χώρα πριν ε, λίγες ώρες ε, το θάνατο της Λουτμίλα Αλεξέβα, η οποία το 2009 έλαβε το βραβείο ε, Ζαχάροφ ως μέλος του Memorial, η Λουτμίλα Αλεξέβα. Εκτός από ότι είχε βραβευτεί από εμά πριν 9 χρόνια, ήταν μία από τις πιο γνωστές ε, αγωνίστριες ε, κατά της ε, Σοβιετικής Ένωσης και ήδη από τη δεκαετία του 70 είχε αγωνιστεί για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα για πάνω από 50 χρόνια. Και το λέω αυτό με αφορμή την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ στον Όλεξ Σέντσοφ φέτος, ο οποίος όπως η Αλεξέβα, όπως και ο ίδιος ο Ζαχάροφ, αποτελεί θύμα του κομμουνισμού. Αυτό που έχουμε τώρα στη Ρωσία αποτελεί συνέπεια ενός πληρούς αποκομμουνισμού. Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί είναι στη φυλακή γιατί δεν έχει πεθάνει δυστυχώς ο κομμουνισμός και ο αγώνας για την ελευθερία σήμερα δίνεται κατά των συνεχιστών. Και αυτό εξηγεί άλλωστε τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας. Εξηγεί το γεγονό ότι ο εύξηνος πόντος δεν είναι μια θάλασσα ελεύθερη. Πολύ συχνά μιλάμε και για τη Μεσόγειο. Επειδή Σήμερα τη διασχίζουν άνθρωποι που επίση ε, θέλουν την ελευθερία. Όμως η Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται υπό αυτή την τεράστια πίεση των Ρώσων. Σήμερα λοιπόν ε, τιμάμε τον κύριο Σέντσοφ με τον πρεβείο Ζαχάροβ γιατί όπως η Αλαξέβα, όπως και πολλοί άλλοι πολίτες από τις ε, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες αγωνίζονταν για την ελευθερία. Δεν έχει τελειώσει αυτός ο αγώνας, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί όσο αυταρχικοί άνθρωποι θα είναι στην εξουσία. Ας ε, τηρήσουμε ζωντανή την ελπίδα μας, λοιπόν, ε, και ε, φυσικά στρέψουμε την προσοχή μας και στη Μεσόγειο, αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Ας διατηρήσουμε το βλέμμα μας υπό τη σκοπιά της ελευθερίας. Σας ευχαριστώ πολύ.